information to all the members of each committee and... Ενημέρωση για όλα τα μέλη ε, της Επιτροπής ε, ε, Μεταφορών και όλων των άλλων συνδεδεμένων επιτροπών. 5 Νοεμβρίου 2018 είναι η επόμενη συνεδρίασή μας, 3 με 6.30 το απόγευμα. Δευτέρα. 5 ε, Νοεμβρίου. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου. Το λέω αυτό για τους συναδέλφους Επιτροπής μας. Περιμένουμε τώρα τους συναδέλφους ε, από την Επιτροπή Μεταφορών. Προσέρχονται. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ από δύο επιτροπές. Καλώς ορίσατε μέλη της Επιτροπής Μεταφορών στην Επιτροπή μας. Εάν ε, δεν έχετε πρόβλημα και παρατηρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Να σας κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, υπάρχει ε, ε, βοήθεια προς τις πολιτικές ομάδες. Έχετε τα έγγραφα μέσω του e-meeting για όλα τα μέλη Ήτρε και Τραν, τους βοηθούς και τις πολιτικές ομάδες κτλ. Εδώ συμπροεδρεύουμε την κυρία Καριμά Ντελή, η οποία συμπροεδρεύει και μαζί με μένα θα είναι και εκείνη υπεύθυνη για αυτή την κοινή μας συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν θέλετε κυρία Ανταλή να πείτε δύο λόγια στην αρχή της συνεδρίασης. Κύριε Μπούζεκ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά και για μένα που βρισκόμαστε εδώ σε αυτήν την ε, κοινή συνάντηση μαζί σας. Αλλά αυτά τα πηγαδάκια και ο θόρυβος που ακούγεται ε, θα ήθελα να σταματήσει γιατί εδώ πρέπει να συγκεντρωθούμε. Μιλάμε για μηχανισμούς, για μηχανισμό διασύνδεσης, μιλάμε για πράγματα πολύ συγκεκριμένα και επομένως πρέπει να έχουμε όλο το μυαλό μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τα μέλη του συναδέλφου της Επιτροπής Μεταφορών, αλλά βεβαίω ε, και τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε για αυτήν την πολύ ανοιχτή ε, και σε βάθος συζήτηση που θα ακολουθήσει. Μιλάμε για έναν ισχυρό μηχανισμό διασύνδεσης που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Ευρώπη και για την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των μεταφορών αλλά και για την μεταφορά ενέργεια ε, για το ψηφιακό και όλα αυτά μέσα, μέσα σε συνθήκες συνέργεια. Όσον αφορά ιδιαίτερα τις μεταφορές, για μα οι στόχοι είναι πολύ σαφεί. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, ε, συνδέουν τους Ευρωπαίους πολίτες, τι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τι δομές και υποδομές και δημιουργούν το απαραίτητο και υπόβαθρο για την μελλοντική κινητικότητα, την κοινωνικότητα του μέλλοντος που θα είναι διασυνδεδεμένη και σύγχρονη. Ε, ε εμείς ε, στρέφουμε το βλέμμα προς το μέλλον, το προετοιμάζουμε και ακριβώς προετοιμάζουμε τις επόμενες δεκαετίες. Θα ήθελα να πω στους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές ότι τους εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτήν την κοινή ε, ε, το κοινό εγχείρημα ε, των δύο επιτροπών και να στεφθεί η, από επιτυχία η προσπάθειά τους και η εργασία τους. Ευχαριστούμε αγαπητή Καριμά, πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες. Υπάρχει ιστορικό συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών, γιατί πριν από 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι και καλά, ε, το πρόγραμμα Connecting Europe Facility είχε αποφασιστεί από δύο ε, και από τις δύο επιτροπές, ε, από την Επιτροπή Μεταφορών και την Επιτροπή Ήτρε. Άρα, ουδέν νέων. Τα γνωρίζουμε αυτά, τα έχουμε ξανακάνει και επί τη βάση του άρθρου 55 έχουμε μοιρασμένη αρμοδιότητα στις δύο επιτροπές. Θα συζητήσουμε λοιπόν το θέμα μαζί και στην επόμενη συνεδρίαση και η ψηφοφορία θα γίνει και στις δύο επιτροπές από κοινού. Να προσθέσω. Έχουμε πάνω από 1.200 ε, τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί διότι βέβαια το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ακριβώς εξηγεί, ε, ε, αυτό δικαιολογεί και τους τρεις εισηγητές. Ο συνάδελφος Μαρινέσκου από είχε Βερκούνεν και ο Πέτρο Τελίτσκα. Έχουμε δύο εισηγητές από τις μεταφορές και έναν από την Ήτρε. Να ξεκινήσω λοιπόν δίνοντας το λόγο στους εισηγητές μας. Ίσως να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία. Κυρία Βιρκούνεν λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, να αρχίσουμε ε, από βιομηχανία και ενέργεια, γιατί οι μεταφορές είναι πιο περίπλοκες και οι περισσότερες δραστηριότητες των κρατών μελών εστιάζουν στις μεταφορές. 1.200 τροπολογίες ακούσατε έχουν κατατεθεί, οι περισσότερες για τις μεταφορές, τα παρατήματα και το Ταμείο Συνοχής. Από πλευράς Ήτρε, ο τομέας ενέργειας και ο ψηφιακός τομέας είναι σαφής. Ε, ο, ο τομέας ενέργειας θα συνεχίσουμε, ε, θα εστιάσουμε στην ενέργεια στα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Ε, θα έχουμε καταγράψει πολύ σημαντικά προγράμματα και το καινούριο στοιχείο, οι ανανεώσιμες και το νέο πρόγραμμα για τις ανανεώσιμες. Η Κομισιόν προτείνει 10% του ενεργειακού project να πάει σε αυτό το τομέα, σε ανανεώσιμες. Πολλά μέλη κατέθεσαν και εδώ τροπολογίες στη νέα πρόταση. Ο ψηφιακός τομέας ίσως δεν είναι τόσο συνεκτικός, γιατί υπάρχουν διάφορες δράσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το ψηφιακό κομμάτι. Προγράμματα, έργα που επιταχύνουν την συνδεσιμότητα σε gigabits ε, και προωθούν κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ε, ε, ασύρματες διασυνδέσεις, μπορούν να χρηματοδοτηθούν επίσης από το πρόγραμμα ΣΕΦ, Μηχανισμό Συνδέοντας στην Ευρώπη, και πολλοί οικονομικές επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ΣΕΦ. Αυτά είναι ξεκάθαρα η ενέργεια, και ο ψηφιακός τομέας. Έχουμε κατάλογο έργων και τομέων ήδη και έχουμε και καλές τροπολογίες από τους ευρωβουλευτές. Ένα σημαντικό θέμα είναι ο προϋπολογισμός, ε, πολύ ενδιαφέρον θέμα από την άποψη του μεγέθους του προϋπολογισμού, από την άποψη του Κοινοβουλίου. Ε, την Άνοιξη το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι το επόμενο πρόγραμμα ΣΕΦ θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος όπως το τρέχον πρόγραμμα και στα ψηφιακά και στην ενέργεια θα πρέπει, είναι ε, το ίδιο όπως το παρόν πρόγραμμα, οπότε εδώ μας ικανοποιούν οι προτάσεις της Κομισιόν. Επίσης, ε, καλό είναι να πούμε το ανέφεραν κι άλλοι, ότι η Κομισιόν προτείνει 60% αυτού του προγράμματος να χρησιμοποιεί δράσεις που συμβάλλουν ε, στη βελτίωση του κλίματος. Γιατί αν χάσουμε ε, στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 25% ε, θα εστιάζονται σε κλιματικές δράσεις. Αυτό το πρόγραμμα είναι όμως στην πρόταση της Κομισιόν 60% για το κλίμα. Όλα τα μέλη θέλω να ευχαριστήσω και για τις 1200 τροπολογίες. Τώρα αρχίσαμε να εργαζόμεθα με τους σκιώδεις και με τους συνεισηγητές, όπως είπε ο Πρόεδρος είναι κοινή η έκθεση αυτή και συνεχώς οι δύο επιτροπές, οι συγητές, οι σκιώδες θα συνεργάζονται. Έχουμε στην ομάδα μας περίπου 20 ανθρώπους, ικανός αριθμός και θα είναι πολύ καλή και η έκθεση που θα σας παρουσιάσουμε, είμαι βεβαία. Ε, κάτι που με λυπεί λιγάκι είναι το εξή. Ξέρουμε ότι στο παρόν πρόγραμμα, στο τρέχον, κάτι που δεν πετύχαμε είναι οι συνέργειες και στην ε, και ενέργεια. Εδώ πρέπει να τα πάμε καλύτερα στο επόμενο πρόγραμμα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε πολύ καλές ιδέες σε αυτό το τομέα, γιατί σχετικά δεν κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες. Κάτι λείπει, υπάρχει μια έλλειψη εδώ. Πρέπει να βρούμε καινούριε ιδέες για να επιταχύνουμε την πρόοδο. Ε, σχετικά με τις συνέργειες, ενέργεια μεταφορές και ψηφιοποίηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αναζωγόνηση των οικονομιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν από την Ήτρε. Τώρα έχουμε δύο εισηγητές από την Επιτροπή Μεταφορών, την Επιτροπή Τρανς, ο συνάδελφος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες σας. Τις ε, εξήτασα όλες ήδη και έχω και ε, ε, σκεφτεί συμβιβαστικές. Οπότε Ήδη έχω κάνει μια αξιολόγηση μέσα από τις συμβαστικές τροπολογίες. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολο να συμφωνηθούν, αλλά δεν είναι πολλά. Υπάρχουν μερικά. Ίσως με ψηφοφορία θα λυθούν, αλλά νομίζω ότι στα περισσότερα θέματα μπορούμε να βρούμε συμφωνία. Τώρα ε, αξιολογούμε τις προτάσεις Αύριο θα είναι η δεύτερη συνάντηση με τους Κιώδης και θα υπάρχει κάτι επιτάπητος ως συμβιβαστικές προτάσεις, κάποια άρθρα. Τώρα για τις μεταφορές, εγώ εργάζομαι άριστα με τον συνάδελφο Πάβελ Τέλιτσκα, οπότε θα καταφέρομαι να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες που θα ικανοποιήσουν όλους τους ε, συναδέλφους. Ένα πράγμα να πω για τον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε μια διαδικασία για το Κοινοβούλιο και πώς θα εργάζεται. Οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Προϋπολογισμού ήδη πρότειναν στην ενδιάμεση έκθεση κάποια νούμερα για όλες τις πολιτικές και αύριο ελπίζω να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Προτείνω να ακολουθήσουμε την πρόταση των εισηγητών, που είναι και συνεισηγητές, εισηγητές για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρόταση είναι να αυξήσουμε τη ε, κονδύλια για τις μεταφορές κατά 7 δις περίπου για να φτάσουμε στην πρόταση της Κομισιόν του 2011, σχεδόν. Βέβαια θα γίνει διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο ε, πάνω στη βάση ελπίζω μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αλλά καλό είναι να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με ένα στιβαρό αίτημα ε, δημοσιονομικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τελίτσικα, πάλι εκ μέρους Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μερικά σχόλια. Θα ήθελα να πω ε, ότι εκτιμώ ιδιαίτερος... Ε, ε, τη συνεισφορά όλων των ε, συναδέλφων με τις τροπολογίες τους. Ε, πολλές νύχτες μείναμε άγρυπνοι διαβάζοντάς τες. Πολλές ήταν πάρα πολύ καλές, πολύ συγκεκριμένες επί της ουσίας. Μερικά σημεία ήταν πραγματικά πάρα πολύ θεμητά και θα τα λάβουμε υπόψη συμβιβαστικέ τροπολογίες από κοινού με τον Μαριάν. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι κάποιες τροπολογίες επαναλαμβάνονταν συνεχώς και πρέπει να αναρωτηθούμε και για την νομική ποιότητα της ε, πρότασης, οπότε θα, προσπαθούμε να, θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε κάπως αυτήν την ε, επανάληψη <clears throat> για λόγους αφήνειας και ποιότητας του κειμένου. οι ιδέες των μόνους, της απλοποίησης ε, των δύο φάσεων και της αξιολόγησης νομίζω έγιναν αποδεκτές σε μεγάλο βαθμό. Φαίνονται, φαίνεται από τις τροπολογίες ε, για τα κριτήρια υπήρξαν περισσότερες τροπολογίες, θα πρέπει να τις ε, διαχειριστούμε και να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε, να δούμε τι πρέπει να υπάρχει σε αυτό το κείμενο και τι αλλού. Το θέμα του προγραμματισμού που προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε με την νομοθετική μας πρωτοβουλία. Ε, μάλλον τα καταφέραμε, τον προϋπολογισμό τον αναφέραμε, οπότε δεν λέω πάρα πολλά, για, δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Το θέμα της κινητικότητας ήταν σημαντικό στην Επιτροπή Μεταφορών κατά την ψηφοφορία και βλέπω ότι υπάρχει υποστήριξη γι' αυτό. Ένα πρόβλημα θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει ένας ε, πληθωρισμός τροπολογιών, μπορώ να το καταλάβω αυτό αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη έμφαση όσον αφορά τους στόχους ε, των Παρισίων, ε, της συμφωνία των Παρισίων το 2020, το καταλαβαίνω, είναι αντιαμφισβήτητο αυτό, αλλά πρέπει να βρούμε την καλύτερη διατύπωση και να δούμε κατά πόσο κάποια στοιχεία έχουν θέσει σε άλλο νομοθέτημα. Για τις περιφέρειες τώρα, ε, που διατρέχουν όλο το πολιτικό φάσμα ε, και που ξεκινούν σε διάφορες ε, ε, περιφέρειες, τα προγράμματα που ξεκινούν σε διάφορες περιφέρειες και διατρέχουν όλο το πολιτικό φάσμα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε βάσει των κριτηρίων ποια πρέπει να κρατήσουμε και ποια όχι. Έχουμε την πλειοψηφία των ε, τροπολογιών που αφορούν ε, την μεταφορά από τα Ταμεία Συνοχής. Ε, μπορούμε λοιπόν να είμαστε απασχολημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό για αυτό το θέμα, αλλά θα το προσπαθήσω. Υπάρχει μία ακόμη συνάντηση σκιωδών αύριο. Θα υποβάλουμε πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες σε αυτήν και θα περιμένουμε τη δική σας συνεισφορά ε, μετά από την συζήτηση αυτή. Πάμε τώρα στους σκιώδεις συζητητές. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη τώρα... Ε, ε, μιλάς εκ μέρους της Ήτρε ή και των δύο ε, επιτροπών. Από την Ήτρε λέει η κυρία Νάτρη. 16 είμαστε και 16 θα παραμείνουμε. Βλέπετε, δουλεύουμε όλοι μαζί. Πολλά άρθρα αφορούν ολόκληρο το πακέτο. Καταρχάς, ε, να πω ότι έλαβα υπόψη ε, τις ε, τροπολογίες σε σχέση με την συνοχή με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και κάποιους γενικούς κανόνες που πρέπει να εγκρίνουμε. για τη συνοχή του ΠΔΠ. Είδα και κάποιες τροπολογίες ε, ε, που φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν ε, που, που, πηγαίνουν προς την κατεύθυνση και των δύο επιτροπών. Εντάξει, δεν υπάρχει ομοφωνία, αλλά είδαμε ότι πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται με την κυρία Βίρκανεν και με τους υπόλοιπους και όδης συζητητές θα προσπαθήσουμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της συνοχής και ε, του ψηφιακής Ευρώπης. Θέλουμε να υπάρξει αποτέλεσμα σε σχέση με τη Συμφωνία των Παρισίων. Μετά από, όλες τις δουλειές που έχω, από όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει για τέσσερα χρόνια, δεν θέλουμε να ξεχάσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Έχουμε νομοθεσία Υπάρχουν ε, οι αγορές ενέργεια στην Ευρώπη ε, και τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη η ενεργειακή αποδοτικότητα. Υπάρχουν πολλά σχόλια γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Αν αφορά τώρα το συνδέοντα στην Ευρώπη, αν έχουμε συνδεδεμένες αγορές ε, ενέργεια στην Ευρώπη, το σημαντικό είναι επίση να λάβουμε υπόψη την αποδοτικότητα και είναι παράλογο να λέμε ότι δεν τη λαμβάνουμε υπόψη ή ότι χρηματοδοτούμε κάτι λιγότερο οικονομικό για να έχουμε ενδεχομένως ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο μέλλον. Ε, πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε μαζί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο, ούτως ή άλλως μέχρι τις 27. Ε, Όπως είπε και η κυρία Βίρκουνεν, υπάρχει το θέμα των διασυνοριακών ανανεωσίμων. είναι όντως ε, σε διασυνοριακό ε, σημείο ή είναι σε, μια, ε, σε ένα σημείο που διευκολύνει τους διαδρόμους για παράδειγμα ακόμη και αν υπάρχει ο διάδρομος, υπάρχει το σιδηροδρομικό δίκτυο ή αυτοκινητόδρομος πρέπει το ίδιο να ισχύει. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε οι μετρητές να υπάρχουν μόνο στους ε, αυτοκινητόδρομους αλλά και στους κόμβους. Ε, δεν θα ήθελα η οι κοινωνικοί κόμβοι ας πούμε να ληφθούν υπόψη τώρα και σε πέντε χρόνια να έχουν ξεχαστεί τελείως. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους κοιόδης να μιλούν το πολύ δύο λεπτά γιατί έχουμε πολύ μεγάλο κατάλογο εισηγητών. Κυρία Γέλα από την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μόλις ε, λάβαμε το έγγραφο δεν μπορέσαμε να τα ε, δούμε. Μια σειρά λοιπόν τροπολογιών συμβιβαστικών ε, που θα συζητηθούν αύριο στην Επιτροπή, στην, συγγνώμη, όσον αφορά τουλάχιστον τις μεταφορές, θα συζητηθούν μεταξύ των σκιωδών και ο κύριος ε, Μαρινέσκο, και η κυρία Τελίσκα, ε, αναφέρθηκαν σε πολλά από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ασχοληθώ μονάχα με θέματα μεταφορών και με θέματα που αφορούν την επιλεξιμότητα και ε, την ε, κυρίως όσον αφορά την πολυτροπικότητα, τα αεροδρόμια, ε, το, την συντήρηση αλλά κυρίως το κύκλο ζωής, την βιωσιμότητα για την μεταφορά εμπορευμάτων δια σιδηροδρόμου, καθώς επίσης και θέματα γεωγραφικής περιφερειακή συνοχή και συνεργασία με τι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, επιλεξιμότητα δράσεων υποστήριξης και βεβαίως εδώ θα υπάρξει ένα άρθρο το οποίο ε, θα προλάβει κατά κάποιο τρόπο την συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Επίσης τροπολογίες οι οποίες ε, σχετίζονται με την ε, διητή κινητικότητα. Κινητικότητα δηλαδή και στρατιωτική και μη στρατιωτική που θα έχει εξειδικευμένο προϋπολογισμό, αλλά εάν δεν χρησιμοποιηθεί 100% ο στρατιωτικός ε, προϋπολογισμός, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να επιστραφεί στις μεταφορές. Αυτό εμείς το υποστηρίζουμε. Επίσης, συμφωνούμε και θα δούμε τι συμβαίνει με την και πώς θα προχωρήσει το θέμα της συνοχής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Έχει να κάνει με το παρελθόν, αλλά εμείς θέλουμε να υπάρχει και μέλλον. Τέλος, να πούμε ότι όσον αφορά τις ε, μελέτες ε, πέρα από την πρόταση ε, μείωσης, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες συμμετέχουν στην βιωσιμότητα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να απαιτήσουν συγχρηματοδότηση σημαντική όσον αφορά το παράρτημα να πω ότι ε, έχουμε κάποια εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά τις, ε, τα, τα, τα διαμεθοριακά, διασυνοριακά, ε, καθώς επίσης και τους νέους δρόμους για το δίκτυο της Βαλτικής και την σύνδεση Βαλένθιας με την Μεσόγειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, συνάδελφο Τσέσακ από την Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Εγώ επικεντρώνομαι σε αυτές που αφορούν βασικά θέματα. Για την ECR είναι σαφές ότι Οποιεςδήποτε μεταφορές από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως για το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Και χαίρομαι διότι ε, το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές υπέβαλαν παρόμοιες τροπολογίες. Ας δούμε δύο έργα που αφορούν τις μεταφορές. Πώς θα ανταγωνιστούν για τη χρηματοδότηση. Πώς θα συγκρίνουμε ε, προγράμματα δύο διαφορετικών κρατών μελών που οι ανάγκες είναι διαφορετικές, οι υποδομές και η ιστορία, οι ιδιαιτερότητες είναι διαφορετικές κάθε φορά. Κάθε κράτος μέλος έχει μια μοναδικότητα όταν πρόκειται για την επέκταση του δικτύου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των κρατών μελών, ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα δεν επαρκούν. Τώρα, όταν πρόκειται για επιλέξιμες δράσεις και τη τροπολογία 97, αυτό που προτείνει η Κομισιόν ε, στην πρότασή της είναι ε, περιοριστικό. Μάλλον, δεν θα περάσει η πρόταση, γιατί είναι πολλοί οι περιορισμοί προκειμένου περιφυσικού αερίου. Οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες και να μας επιτρέψουν να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, να μπορέσουμε να προωθήσουμε εναλλακτικά καύσιμα και να βελτιώσουμε τη ρήπανση του αέρα. Μπορούμε έτσι να προωθήσουμε ανανεώσιμες πηγές. Όλα έχουν να κάνουν με τις τοπικές συνθήκες και με το τοπικό ενεργειακό μείγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην Άλντε. Μόρτεν Χέλβεκ Πέτερσεν δεν είναι εδώ ο σκιώδης της Άλντε. Εξ του Μόρτεν και η κυρία Τέλιτσκα, ο κύριος Τέλιτσκα. Τώρα θα βάλω το καπέλο της Σίτρε. Ε, ζητώ συγγνώμη για τον Μόρτεν που είχε άλλες υποχρεώσεις. Μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω και ο Μόρτεν θέλει να πει ότι θέλει να εκφράσει την εκτίμησή του στους συζητητές για την καλή εργασία στην έκθεση αυτή ε, το ΣΕΦ είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Η IPCC έκθεση κάνει μια ανησυχητική παρατήρηση ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλή δουλειά για τα κλιματικά και τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το ΣΕΦ, το μηχανισμό, ε, ως δυνατότητα να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις και να μειώσουμε τις ε, εκπομπές. Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη το Κοινοβούλιο να είναι ενωμένο στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν. Θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να ε, προσβάλλουμε το ε, status quo και το Συμβούλιο όταν στυλώνει τα πόδια όταν πρόκειται για την ενεργειακή μετάβαση. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Από την Γκουε. Η Σκιώδης εκπροσωπούνται και οι δύο επιτροπές εκπροσωπούνται από την Τάνια Γκοντζάλες Πένιας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους τρεις εισηγητές για την οργάνωση αυτής της συζήτησης. Θα μιλήσω εξ ονόματός μου ε, για την Επιτροπή Μεταφορών, αλλά επίσης και εξ ονόματος ε, του συναδέλφου Χαβιέρ Μπενίτο, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ και ζητά συγγνώμη, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και θα, θα πω μερικά λόγια ε, για εξ ονόματός του όσον αφορά την εργασία του για την Επιτροπή Ήτρε. Ε, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Μας, ε, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, η αρχή της ενεργειακής αποδοτικότητας να αποτελέσει οδηγό και θα πρέπει πριν δούμε οι υποδομές να δούμε με ποιο τρόπο θα αποφύγουμε την δημιουργία νέων υποδομών ε, που ενδεχομένως δεν θα ε, είναι ανάλογες με τις ανάγκες. Επίσης θα πρέπει να σταματήσουν ε, ή ε, οποιασδήποτε επενδύσεις σε, ορυκτές, ε, σε ορυκτά καύσιμα συμπεριλαμβανομένου και του λεγόμενου φυσικού αερίου και οπωσδήποτε να ληφθούν τα μέτρα αυτά τα οποία θα μας προσαρμόσουν στη συνθήκη και τη συμφωνία των Παρισίων. Να πω ότι έχουμε πάνω από 1.200 τροπολογίες και λίγο χρόνο και επομένως ενδεχομένως θα είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ ε, του μείγματος αλλά παρόλα αυτά μας ενδιαφέρει να έχουμε καθαρό ε, και ε, σύγχρονο σύστημα μεταφορών. Στις τροπολογίες μου προσπάθησα να θέσω κάποια ζητήματα ας πούμε να μην μείνουν εκτός επιλεξιμότητας ε, το ε, τμήμα ε, που συνδέει την Βαλένθια, τη Σαραγώσα και φτάνει μέχρι, περνάει από τον Ατλαντικό, εν πάση περιπτώσει στην Μεσόγειο, περνώντας από την ε, από την Καντάβρια ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να έχουμε και τις απαραίτητες νομοθετικές διοικητικές ρυθμίσεις για οποιαδήποτε νομοθεσία προχωρούμε. Επίσης το θέμα και η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας είναι σημαντική. Εγώ δεν λέω, δεν αμφισβητώ ότι το φυσικό αέριο δεν είναι λίγο πιο καθαρό από το πετρέλαιο πετρέλαιο αλλά δεν, είναι, ε, δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι ε, όσον αφορά την μία ή την άλλη πηγή ενέργειας γιατί πιστεύω ότι εδώ πέφτουμε σε μία παγίδα ε, γιατί τελικά οι καθαρές μορφές ενέργειας και η μείωση των εκπομπών είναι το πιο σημαντικό. Ναι, τελειώνω, τελειώνω, είμαι πολύ σύντομη παρότι μιλάω εξ δύο ανθρώπων. Ε, επίσης ε, θα πρέπει οπωσδήποτε 100% ε, προσβασιμότητα να έχουν σε ανθρώπους με αναπηρία όλες οι υποδομές οι, δημόσια, οι δημόσιες μεταφορές θα είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να προηγηθούν και είναι αυτές οι οποίες θα μας επιτρέψουν να είμαστε εγκύτεροι προς τους πολίτες και να τους βοηθήσουμε πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Γκονσάλες Πένιας. Έχετε δίκιο, γιατί ε, μιλάτε εξ ονόματος δύο, έχετε το χρόνο δηλαδή δύο ε, εισηγητών. Εξ ονόματος των Πρασίνων θα δώσω το λόγο στον Μίχαλ Κράμερ από την πλευρά των μεταφορών. Όχι, δεν είναι εδώ, αλλά η Πρόεδρος θα τον αντικαταστήσει. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, εξ ονόματος του κυρίου Μίχαελ Κράμερ έχω να πω τα εξή. Οι μηχανισμοί διασύνδεσης θα πρέπει να ξαναβρούν τους κεντρικούς άξονες. Η κινητικότητα του μέλλοντος θα πρέπει να συνδυαστεί με το θέμα της εγκύτητας ε, έτσι ώστε να σταματήσουν τα μεγάλα ανώφελα προγράμματα. Ε, ξέρετε, ας πούμε, το θέμα του ε, Ρήνου που απασχολεί πολύ τον κύριο Κράμερ. Δεύτερον, ε, τον 21ο αιώνα το σημαντικό δεν είναι να οικοδομήσουμε και ακόμα και περισσότερα και περισσότερες ε, ε, υποδομές, αλλά να γίνει ανανέωση όσον αφορά το σιδηρόδρομο, όσον αφορά τους οδικούς άξονες. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, κλειδί του 21ου αιώνα είναι η διατροπικότητα ή η πολυτροπικότητα και πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την πολυτροπικότητα και η, ιδέα που πρέπει να μας ε, ε, οδηγεί είναι ότι 70% ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και των ε, που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αφορούν 70% λέω προέρχονται από τις χερσαίες μεταφορές. Απ' την άλλη πλευρά έχουν, αυξάνονται διαρκώς τα, φαινό, ε, οι εκπομπές που οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, επομένω όλοι οι τομείς θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και επομένως ε, η ηλεκτρική ενέργεια ε, που θα προέρχεται από αναγενεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο αλλά και υδρογόνο. Τέλος, η κινητικότητα της αυριανής μέρας δεν μπορεί να είναι πραγματικά κινητικότητα του, 21ου αιώνα εάν δεν είναι προσβάσιμη σε όλους. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους ε, που έχουν μεγάλη επισφάλεια όσον αφορά την ε, κινητικότητα, κυρίως ε, στις περιοχές της Υπέθρου. Αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στους μελλοντικούς μηχανισμούς διασύνδεσης. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και από την Επιτροπή Ήτρε ο συνάδελφος Μαρτσελέζη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι, ε, ότι δεν ε, υπάρχουν πλέον ε, αμφιβολίες μετά από την χθεσινή παρουσίαση στα Ηνωμένα Έθνη της ε, ε μελέτης εγκρίτων επιστημόνων και έχουμε ε, από την άλλη πλευρά ε, πολλά εκατομμύρια θέσεων εργασίας ε, που μπορούν να δημιουργηθούν. Με το ΣΕΦ μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εάν με προϋπόθεση όμως να μην βάλουμε ούτε ένα ευρώ πλέον στα ορυκτά καύσιμα και γι' αυτό λοιπόν τον στόχο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην βάλει ούτε ένα ευρώ στα green συστάσεις. Επίσης, 70% των ε, προγραμμάτων ε, θα πρέπει να, τους θα πρέπει να αφορούν το κλίμα. Επίσης, climate proofing ζητούμε διασυνοριακά προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Κομισιόν έδωσε ένα 10%, την ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό. Ε, θέλουμε τουλάχιστον 20%, τουλάχιστον λέω. Τέλος, ε, επανέρχομαι στην αρχή ε, της ενεργειακής ε, ένδυας. Δεν θα πρέπει ε, να βρούμε, να εφεύρουμε κάτι καινούριο. Έχουμε ήδη την ασφάλεια, το κείμενο για την ασφάλεια της προμήθειας αερίου. Έχουμε επίσης αυτή, αυτό το κείμενο το οποίο δεν λέει ότι θα επενδύσουμε καινούρια χρήματα σε νέα προγράμματα, αλλά θα δούμε εάν υπάρχει η δυνατότητα ε, σε παλιά προγράμματα να επιτευχθεί η ε, ενεργειακή αποταμίευση. Νομίζω ότι ε, έχει ήδη ακουστεί ο κόδωνας του κινδύνου και θα πρέπει τώρα να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να περάσουμε στην οικολογική μετάβαση. Ευχαριστώ. Σκιώδης εισηγητές από την EFTD. Ταμπουράνο και για τις δύο επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις τροπολογίας ε, δικές μας ε, που αφορούν ε, ψηφιακές ε, υποδομές και μετά θα πω δύο λόγια για την Επιτροπή Μεταφορών. Εμάς μας ενδιαφέρει η αντοχή απέναντι στην κλιματική αλλαγή, η πλήρης απανθρακοποίηση ε, της ε, οικονομίας ε, και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Connecting Europe Facility να έχουν το climate proofing καθώς επίσης και να είναι ανθεκτικά όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσουμε σε νέες υποδομές ε, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω σε οτιδήποτε σχετίζεται με ορυκτά καύσιμα, ακόμα και με το φυσικό αέριο. Η αντίληψη ε, ότι πρώτα θα πρέπει να μας απασχολήσει η ενεργειακή αποδοτικότητα. Εδώ ε, δεν ε, σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαδεθούν τα προγράμματα σε διασυνοριακά προγράμματα, έστω και αν αυτά παρουσιάζουν μεγάλη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Λέμε όμως ότι πριν χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα ε, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες και οι δυνατότητες μείωσης της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό είναι πολιτική απόφαση και διαθεσμική ε, απόφαση. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να μην λησμονούμε σε καμία περίπτωση την ηλεκτρομαγνητική ρήπανση η οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για διασυνδεσιμότητα και για τεχνολογίες των οποίων την επικίνδυνοτητα δεν γνωρίζουμε ακόμα κυρίως όταν εγκαθίστανται ε, κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Η πρότασή μας να ε, ε, έχουμε πιο ασφαλείς ε, και σίγουρες υποδομές εστιάζεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε, να έχουμε μάλλον ευαισθησία όσον αφορά την καθημερινότητα και την καθημερινή ζωή των πολιτών και να μην έχουμε σαν κύριο γνώμονα μονάχα την αγορά και το κέρδος πολλές ε, ε, οι υποδομές πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουν ασφάλεια και επομένως ε, δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μονάχα την Ιταλία. Εμείς ε, λέμε ε, ότι το ΣΕΦ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για νέες δομές μεταφορών αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση και ενημέρωση των και επικαιροποίηση των υπαρχουσών υποδομών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Ντάριο. Η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας επίσης ε, γνωμοδοτεί. Μάσιμο Καστάλντο είναι ο εισηγητής. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Είστε ο συντάκτης γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας λέω ότι παρότι είχαμε λίγο χρόνο ε, και με την ε, ε, γρήγορη επιτεχημένη διαδικασία και λόγω του καλοκαιριού είχαμε προβλήματα, παρόλα αυτά καταφέραμε να κάνουμε μια καλή δουλειά. Η υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ προσπάθησε να έχει επαφές με όλες τις ομάδες. Ευχαριστώ τους Χιώδης και τη Γραμματεία γι' αυτό. Θέλουμε να στείλουμε σαφές ε, μήνυμα στις ε, δύο αρμόδιες καθήλοι επιτροπέ ε, επιτροπές έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα διακυβεύματα και οι προκλήσεις όσον αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα. Τέσσερα είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν χαρακτήσει τη δουλειά μας όσον αφορά την στρατιωτική κινητικότητα. Πρώτον, ε, η dual use. Ε, η στρατιωτική κινητικότητα βασίζεται σε συγκεκριμένες μη στρατιωτικές υποδομές. Πρόεδρος, μήπως μπορώ να σας ζητήσω να μην τρέχετε τόσο γιατί ε, α, είσαστε σε αυτοκινητόδρομο μεγάλης ταχύτητας. Έλεγα λοιπόν, λέει ο κύριος Καστάλτο, ότι, θέλουμε, ότι ε, πρέπει οπωσδήποτε ε, οι υποδομές αυτές να μπορούν να διαχειριστούν ξεκινήσουν υλικό ε, και στρατιωτικό και μη στρατιωτικό. Δεύτερο ε, είναι το σενάριο ε, το εξή. Είναι προφανέ ότι η στρατηγική κινητικότητα οπωσδήποτε θα, είναι υπέ, θα, θα, θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Δεν πρέπει να λησμονούμε τις, ε, ε, τα, θέματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια ε, των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν έλλειψη δογματισμού και ισορροπημένη γεωγραφική αντιμετώπιση της στρατηγικής κινητικότητας. Ε, τα σενάρια για τα Βαλκάνια, για την Βόρεια Αφρική, καθώς επίσης και για τον Βόρειο Κύκλο, είναι σενάρια τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν. Ε, Οπωσδήποτε θα πρέπει να προκύψουν και ε, οι συνέργειες με τα προγράμματα του ΝΑΤΟ. Τρίτον, ε, η στρατιωτική κινητικότητα ε, δεν αφορά μονάχα την μετακίνηση δυνατοτήτων και προσωπικού σε περίπτωση κρίσης, αλλά ε, σε περίπτωση ασκήσεων, σε περίπτωση συντήρησης, όπως ας πούμε και σε περίπτωση αντίδρασης σε φυσικές ε, καταστροφές, ε, η κινητικότητά τους, λέω, πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, καθώς επίσης να διευκολυνθούν και όλες οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν διπλωματικές και διοικητικές γραφειοκρατικές διευκολύνσεις. Τέταρτο σημείο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι η περιβαλλοντική διάσταση και η βιωσιμότητα αυτή της στρατηγικής κινητικότητα. σε σχέση δηλαδή με τις εκπομπές καθώς επίσης και σε σχέση με τα υψηλά και επικαιροποιημένα ε, ε, πρότυπα. Εμείς έχουμε ε, έναν αριθμό τροπολογιών που αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία εντός της νομοθεσίας. Επιστεύουμε ότι εάν, έχουμε, αν γίνουν δεκτές οι τροπολογίες μας, οπωσδήποτε θα έχουμε μια ισορροπημένη εκπροσώπηση της υποεπιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να παραχωρήσω την Προεδρία στην κυρία Ντελή. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσει τώρα η συζήτηση για τους ευρωβουλευτές που θα ήθελα να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Πασκουάλ Ντεγκράντε. Έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία του ΕΛΚ ε, θεωρεί ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, για την ε, Ισπανία. Εμείς πλέον είμαστε στην αντιπολίτευση στη χώρα μου, ωστόσο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υπερψηφίσουμε τροπολογίες της σοσιαλίστες συναδέλφου. Το θέμα των μεταφορών ε, έχουμε την τροπολογία 1120 ε, ε, σε σχέση με τη διασύνδεση Σαραγώσα-Βαλένθια, Μαδρίτης μέχρι την Μεσόγειο. Επίσης, Έχουμε την 240, 202 και 1070 που έχει υποβάλει και η κυρία Ντελκαστίγιο. Σημαντικές επίσης όσον αφορά τις αεροπορικές ε, ε, υποδομές. Δεν έχει δώσει και στους αερολιμένες δεν έχει Ε, δεν έχει δώσει προτεραιότητα στα θέματα αυτά. Επίση, τροπολογίε 676, 690, 693, οι οποίε αφορούν τη συγχρηματοδότηση καθώς επίσης και άλλες τροπολογίες ε, δικές μου που αφορούν ε, τις ε, ιδιαίτερα περιφερειακές περιφέρειες κλπ. Υπάρχουν επίσης για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές τροπολογίες οι οποίες αφορούν την απομόνωση και τις... Και τέλος, θα ήθελα να απορρίψω την τροπολογία 957. Θεωρούμε ότι δεν δείχνει μεγάλη αλληλεγγύη η τροπολογία αυτή και επομένως θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και αλληλέγγυοι με το σύνολο της Ισπανίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ με την τροπολογία σας 1120. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του συναδέλφους ε, ε, που, τις τροπολογίες που θέλουν να προωθήσουν τους κόμβους δεν πρέπει μόνο στα διασυνοριακά προγράμματα να επικεντρωθούμε, αλλά αυτοί οι αστικοί κόμβοι να υπάρχουν στην συνέχεια των μεταφορών. Τροπολογία 818 που έχω συνυπογράψει με πολλούς συναδέλφους, αμοιβαιότητα στις δημόσιες ε, ε, προμήθειες ε, για, για την ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιοποίηση γιατί δίνεται η δυνατότητα στις αρχές που αποφασίζουν να ε, μη δώσουν μία προμήθεια σε μία χώρα η οποία δεν έχει συνυπογράψει υπό ίσους όρους μία προμήθεια όπως θα γινόταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει δηλαδή μία συγκρίσιμη ε, πρόσβαση στην ε, δημόσια προμήθεια. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο σχετικό και δίνει τη δυνατότητα αν ένας μηχανισμός διασύνδεσης υποστηρίζει ένα πρόγραμμα αυτό να σέβεται την αρχή της αμοιβαιότητας. Αυτό προωθεί όχι μόνο την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά ε, και την αρχή της αμοιβαιότητας που πάντοτε υπερασπιζόμασταν. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριλάβουμε αυτή την τροπολογία γιατί αν η Επιτροπή απέριπτε κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση στην Ολομέλεια γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να, να ανοίγουμε εμεί τι αγορέ μα σε ανταγωνιστέ όταν οι ανταγωνιστέ κλείνουν τι αγορέ σε εμά. Κύριε Ρικέ, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, δημοσιονομικής ε, φύσεως η παρατήρησή μου, ο μηχανισμός ε, ε, λειτουργήσε πολύ καλά 500 δισεκατομμύρια πρέπει να ε, δώσουμε για να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα όπως πρέπει. Ε, επίσης, ε, στο πλαίσιο των πιστώσεων ΦΕΝΤΕΡ, ανταγωνιστικότητα τουλάχιστον κατά μέσο όρο 70 δισεκατομμύρια έχουν αξιοποιηθεί, αλλά για έργα μεταφορών που δεν έχουν καμία ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όπως δείχνει ο απολογισμός των τελευταίων 15 ετών. Γι' αυτό πρότεινα μία τροπολογία 20 δις ε, ε, απλώς θα μεταφέρει τα 20 δισεκατομμύρια από το ΦΕΝΤΕΡ για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια διαχείριση που είναι ε, κεντροποιημένη και αποτελεσματική και έχει προστιθέμενη αξία. 8% του προπολογισμού του ΦΕΝΤΕΡ είναι. Αν σκεφτούμε ότι 10 δις ε, πήραμε από τα, 4, από τα 40 δις που είχαν προβλεφθεί. Νομίζω ότι είναι μάλλον μετριοπαθές. Αν δεν καταφέρνουμε ένα τμήμα του βετέρ να το μεταφέρουμε σε έναν κεντρικό μηχανισμό, δεν υπάρχει περίπτωση να, να πλησιάσουμε, όχι να υλοποιήσουμε ε, τις, ε, τους στόχους μας για, το, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Λουκαζένσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το συνδέοντα στην Ευρώπη έχει ε, επεκταθεί ε, για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Επίσης συμφωνώ ότι ε, όταν γίνεται προγραμματισμός νέων υποδομών και νέων επενδύσεων πρέπει να χρησιμοποιούμε την κοινή λογική. Τα διασυνοριακά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ, η Επιτροπή Μεταφορών. Πάντοτε ήταν υπέρ του διασυνοριακού εμπορίου με την Ουκρανία. Όμως ε, ο διάδρομος ε, Βαλτικής θάλασσας και Βόρειας θάλασσας τελειώνει στο Κατόβιτσε. Ε, αυτό με προβληματίζει κάπως. Θα έπρεπε να επεκταθεί ε, σε μια, στο Τσέσουφ στην Πολωνία, κοντά στα Καρπάθια, μέχρι το Ουκρανικό σύνορο. Ο διάδρομος 8 ε, θα επεκταθεί, συνεπώς χρειάζεται να υπάρχει μία συνέργεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και όλους τους κυριώδεις εισηγητές γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα και ελπίζω ότι θα είναι, κα, θα είναι καλός ο συμβιβασμός που θα προκύψει και που θα είναι αποδεκτός και από τις δύο επιτροπές. Κάτι ακόμη μικρό να πω. Κάποιες ε, αμφιβολίες έχω σε σχέση με αυτή την κλίδα κατανομής. 70% αντιστοιχεί στα εθνικά ε, ε, ποσά και ε, 30% για όλες τις, τις χώρες πολιτικής συνοχής. 70-30. Αυτή είναι η σωστή κατανομή. Ανησυχώ κάπως γιατί πιστεύω ότι οι μικρότερες περιφέρειες θα καθυστερήσουν και δεν θα μπορέσουν να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις. Ελπίζω να ληφθεί υπόψη αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Λουκασένσκα. Δεν είδα άλλους ε, συναδέλφους να θέλουν να πάρουν το λόγο. Οπότε για να συνοψίσω θα ξαναδώσω το λόγο για ένα λεπτό ε, στους συζητητές μας. Κυρία Βυρκίνεν, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Να ευχαριστήσω όλους σας ε, για τις παρεμβάσεις σας και βεβαίως για τις τροπολογίες. Και όπως είπε και ο Μαρίν Μαρινέσκο, αύριο θα συναντηθούμε με τις Κιώδης το πρωί και θα συνεχίσουμε την εργασία μας. 22 ε, Νοεμβρίου πρέπει να ψηφίσουμε. Οπότε πρέπει να κάνουμε μερικές ακόμη συναντήσεις και γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ενεργό σας ε, συμμετοχή. Κύριε Μαρινέσκου, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Θα λάβουμε υπόψη όλες τις προτάσεις. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ. Ήσασταν σύντομος και ακριβής, όπως πάντοτε. Κύριε Τερλίτσκα, Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ να συμφωνήσω με αυτά. Μας προκαλείτε κύριε Τελίτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς που σας γνωρίζω. Πριν ολοκληρώσουμε, το είπατε κυρία Βρικάνεν, 22 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία, μην φύγετε αμέσω. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, ο μηχανισμός διασύνδεσης Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε το στόχο και τη φιλοδοξία να βρούμε συμβιβασμούς και με την Επιτροπή των Μεταφορών και με την, με την Επιτροπή Ήτρε. Δύσκολο καθήκον. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε για να κάνει και εκείνος κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Αυτά. Ευχαριστώ. Πέρα στη σας. Great. Okay.